I'm going to start on the blue growth. I'll, I'll start with the blue. Θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε την ε, μπλε ανάπτυξη. Γιατί έχουμε και τον εισηγητή. Γαλάζια ανάπτυξη, κύριε Δανέλη. Floor Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι εχθροί της γαλάζιας ανάπτυξης επιχείρησαν να μας αποδυναμώσουν και γι' αυτό δημιούργησαν αυτό το false fire alarm. Εμείς όμως ε, θα επιμείνουμε. Ε, νομίζω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έχει γίνει τόσο πολλής λόγος για την αναγκαιότητα δημιουργίας συνθήκων ενδυνάμωσης της ανάπτυξης, δημιουργίας συνθήκων αναθέρμανσης της πραγματικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει τόσο εφιαλτικά το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας να απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την μπλε ανάπτυξη είναι μια εξαιρετικά φιλόδοξη, οραματική, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική πρόταση για την ε, αξιοποίηση της θαλάσσιας οικονομίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ε, σε πάρα πολλούς τομείς για την πραγματική ανάπτυξη και βεβαίως δημιουργία ε, εξαιρετικά σοβαρού αριθμού θέσεων εργασίας και μάλιστα σε ένα πολύ γρήγορα, γρήγορο και άμεσο χρονικό ορίζοντα. Νομίζω επίσης ότι η στροφή στη θάλασσα πράγμα που είναι γνωστό στην Ευρώπη τα τουλάχιστον 4 με 5.000 τελευταία χρόνια, δίνει μια ευκαιρία στην Ευρώπη να ξανααποκτήσει ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις ε, μεγάλες αναπτυσσόμενες, αναδιόμενες οικονομίες της Ανατολής και του Νότου. Πιστεύουμε ότι βασικά ε, κλειδιά στην ε, επέκταση της γαλάζιας ανάπτυξης στους τομείς ε, τους οικονομικούς τους οποίους αναφέρεται, μας δίνουν οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, θεωρώντας ότι είναι αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση του αυξανόμενου συνεχώς αριθμού των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρούμε στην έκθεσή μας ότι ένας βασικός τομέας ε, που θα πρέπει άμεσα με συγκεκριμένα μέτρα να στηρίξουμε είναι η δημιουργία των ε, ειδικών δεξιοτήτων για την απασχόληση που θα ε, δημιουργηθεί ως ευκαιρία. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ γρήγορα έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα εργατικό δυναμικό που να μπορεί να αξιοποιήσει τις θέσεις εργασίας οι οποίες πολύ γρήγορα θα δοθούν από την ανάπτυξη των τομέων αυτών και γι' αυτό το λόγο νομίζουμε ότι θα πρέπει να συσταθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο, ένα, μάλλον ευρωπαϊκά τομεακά συμβούλια για την απασχόληση και τις δεξιότητες, προκειμένου να καταγραφούν οι νέες τάσεις όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες και κατάρτιση, να υποστηριχθούν προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο για την εκτίμηση των αναγκών σε επαγγελματικέ δεξιότητες και τη διασφάλιση της ενημέρωσης των στοιχείων που περιέχονται στο πανόραμα δεξιοτήτων ΕΕ, όπως επίσης και να ληφθούν πρωτοβουλίες επιμόρφωσης που προωθούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, όπως μια πολιετής δράση για την ανταλλαγή σπουδαστών, καθηγητών και νέων επαγγελματιών τύπου Εράσμους. Σχετικά με την ναυτιλία και την ναυπηγική βιομηχανία, νομίζουμε ότι η πρόθεση των θαλασσίων μεταφορών συμβάλλει όχι μονάχα στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά συμβάλλει και στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Λευκή Βίβλος για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, ώστε να μετατοπιστεί το 50% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στις σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές μέχρι το 2050. Σημειώνουμε με ανησυχία στην εκθεσή μας ότι η ναυτιλία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνεται από υπερβολικές διοικητικές και τελωνιακές διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο το όραμα ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών και γι' αυτό το λόγο μιας και το πιλωτικό πρόγραμμα Γαλάζια Ζώνη είχε ιδιαίτερη επιτυχία, καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία της «Γαλάζια ζώνης ε, εντός του 2013. Επίσης, επισημαίνουμε ότι ο τομέας της ναυπηγικής βιομηχανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πλήττεται ε, τα τελευταία χρόνια ε, εξαιρετικά έντονα, έχει τη δυνατότητα μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης να αυξήσει τη συμβολή του στην ανάπτυξη και απασχόληση με την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που προκύπτουν από τη ζήτηση για τα καθαρά πλοία αλλά και για, την, ε, για τα πλοία τα καινούργια που θα απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Έτσι, εδώ θέλω να επισημάνω ότι θεωρούμε ότι η, η μπλε ανάπτυξη, η γαλάζια ανάπτυξη δεν αναφέρεται μονάχα στις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες της Ένωσης, αλλά αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες του συνόλου της ε, επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό που βεβαίως είναι ίσως η βασικότερος τομέας ε, της μπλε ανάπτυξης και αυτός που άμεσα μπορεί να ενισχυθεί. Εδώ καλούμε τα κράτη-μέλη με την άμεση συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών να στηρίξουν πρωτοβουλίες ανάπτυξη και αναβάθμισης τουριστικών υποδομών και βεβαίως να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εκλείψουν φαινόμενα γραφειοκρατίας και διαφάνειας που πλήττουν σήμερα τον κλάδο. Και θεωρούμε ότι είναι υψίστης σημασίας ο ρόλος των περιφερειακών αρχών στην δημιουργία ή αναβάθμιση εξειδικευμένων σχολών υψηλού επίπεδου διοίκηση και οικονομία τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών επαγγελμάτων, ναυτικών σχολών, σχολών μαγείρων κτλ. Είναι άμεση ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίε των θεωρήσεων, τη έκδοση των θεωρήσεων. Αυτό το λέμε σε κάθε ευκαιρία όταν συζητάμε για τον τουρισμό. Ε, η μείωση του κόστου, η μείωση του χρόνου που απαιτείται, η απλοποίηση των διαδικασιών και η υιοθέτηση έξυπνων τρόπων ε, χορήγηση τουριστικών θεωρήσεων θα μεγιστοποιήσει το εισερχόμενο ρεύμα, κυρίως από τις χώρες BRICS που ε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ο τομέας της κουραζιέρας είναι ένα σημαντικό, ε, μπορεί να παρέχει ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για τα ευρωπαϊκά λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες που τα περιβάλλουν. Ε, μπορεί να ενθαρρύνει το σχεδιασμό ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην επάυξη της εμπειρίας των επισκεπτών δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική και ιστορική σημασία των λιμενικών προϊσμών, δημιουργώντας έτσι μια προστιθέμενη αξία στον τομέα της κουραζιέρας. Ε, ζητούμε από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιμένων μέσω της υποστήριξης λιμενικών υποδομών, αναβάθμισης προσφερωμένων υπηρεσιών, όπως παραδείγματος χάρη την προσαρμογή στις απαιτήσει του Σέγγεν, ώστε τα ευρωπαϊκά λιμάνια να καταστούν ελκυστικότερα για την κουραζιέρα και βεβαίως εποφελέστερα για τις τοπικές κοινωνίες. Υπογραμμίζουμε τη σημασία του κλάδου των σκαφών αναψυχής, yachting, για το θαλάσσιο τουρισμό. Στη Μεσόγειο έχουμε τη μεγαλύτερη αξιοποίηση αυτού του, αυτού του τομέα ε, θαλάσσιου τουρισμού. Καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει στα πλαίσια της μελλοντική ανακοίνωσης για το θαλάσσιο τουρισμό τις δυνατότητες της απλοποίησης και της εναρμόνισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των κανόνων για την έκδοση αδειών λειτουργία, απαιτήσει ασφάλεια, συντήρηση και επισκευή σκαφών αναψυχή, αλλά και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του κλάδου, πράγμα που σήμερα δεν ισχύει. Επίσης, θεωρούμε ότι ο ρόλος της γαστρονομίας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού παράκτηου τουρισμού και όχι μόνο, είναι εξαιρετικά σημαντικός και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ενθάρρυνση των συνεργειών μεταξύ του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής δηλαδή των τοπικών αγροτικών προϊόντων και της σύνδεσης με τον τριτογενή τομέα του τουρισμού ε, δίνει εξαιρετικά ωφέλη όχι μονάχα στις παράκτιες περιοχές της Ένωσης αλλά και στην ενδοχώρα αυτής και εμπλέκει ένα μεγάλο αριθμό ωφελουμένων. Σχετικά με τον τομέα της γαλάζιας ενέργειας, η γαλάζια ενέργεια θεωρούμε όλοι ότι αποτελεί ένα κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή θαλάσσια οικονομία και θα πρέπει η Επιτροπή να στηρίξει ενεργά την παγκόσμια πρωτοπορία που σήμερα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω σε ερευνητικό τομέα, ώστε να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανία στρατηγικής για την καλάζια ενέργεια, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με άλλους κλάδους. Επισημαίνουμε επίσης ότι η, η δημιουργία υπεράκτιων ε, θαλάσσιων ε, ενεργειακών πάρκων θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που σήμερα ε, υπάρχει σε πολλές από τις παράκτιες περιοχές σε σχέση με την ασυμβατότητα δραστηριοτήτων όπως είναι ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, και αυτό θα μπορεί να συνδυαστεί με την δημιουργία πάρκων υδατοκαλλιέργειας που είναι ο άλλος τομέας, βασικός τομέας ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας που ο συνδυασμός και η συνύπαρξη ε, εγκαταστάσεων γαλάζιας ενέργειας υπεράκτιων με, ε, με, με, με υδατοκαλλιέργεια υπεράκτια θα μπορέσει να λύσει επίσης προβλήματα έντασης που δημιουργούνται από τις υπερεντατικές υδατοκαλλιέργειες σε παράκτια οικοσυστήματα και σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισμός που λέγαμε και πριν. Να σημειώσω εδώ ότι ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών στην Ένωση παρέχει ήδη 80.000 θέσεις εργασίας και να σημειώσουμε ότι η εκτίμηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η παραγωγή των εκτρεφωμένων ψαριών θα υπερβεί εκείνη των συμβατικών αλλιευμάτων το 19, το 2019 ε, δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες ε, σε ε, ανάγκης αξιοποίησης των στοιχείων αυτών για την ανάπτυξη των για τον τομέα της θαλάσσιας εξόριξης ορυκτών, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ε, θαλάσσια εξόριξη, όμως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόριξης του θαλάσσιου βυθού. Τέλος, στον τομέα της γαλάζιας βιοτεχνολογίας ε, μπορούν να δημιουργηθούν πολύ γρήγορα θέσεις απασχόλησης ψηλής εξειδίκευσης και βεβαίως προσφέρει ο τομέας αυτό σε κρίσιμου τομείς ήδη με πολύ μεγάλες και εξαιρετικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον σε τομείς όπως η υγεία, η κοσμετολογία, η διατροφή και η καινοτομία. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις για την στενή συνεργασία που είχαμε ε, μέχρι σήμερα και βεβαίως για αυτήν που θα έχουμε και στο επόμενο στάδιο, όπως επίσης ε, τη Γραμματεία και τους συνεργάτες του γραφείου μου για την σημαντικότητα της συμβολή τους στην επίτευξη αυτής της δουλειάς και είμαι στη διάθεσή σας για, τις, ε, για τη συζήτηση την περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βλαστό έχει το λόγο τώρα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα Ευχαριστώ πολύ τον συναδελφό μας τον Σπύρο για το έργο του. Γιατί συμμερίζομαι πολλές από τις παρατηρήσεις που κάνει και πολλές από τις προτάσεις του. Όμως νομίζω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί παρετέρω. Συγγνώμη που το λέω αποτελεί έναν χάρτη πορεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ενισχύσει αυτήν την γαλάζια ανάπτυξη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το, την προστασία του περιβάλλοντος επίσης Κάτι το οποίο ε, μου επιτρέπει να φτάσω στο ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά για να διαρθρώσουμε καλά τα διάφορα εργαλεία για την γαλάζια ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας και τις υπάρχουσες στρατηγικές αλλά και τις μελλοντικέ που θα υπάρξουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι συμφωνούμε για το ότι πρέπει να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το ε, ίχνος του άνθρακα, τέλο πάντων της ρήπασης της ατμόσφαιρας και στις παράκτιες περιοχές. Να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές, εννοείται πρέπει να το φροντίσουμε αυτό και η έκθεση αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται κάποιο παρετέρω διευκρίνηση. Έχω και κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, να κάνω. Στηρίζω την ιδέα ότι χρειάζεται ευελιξία στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων ε, γραμμών από τα κράτη-μέλη αυτές που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε να μπορούν να τις θέσουν σε εφαρμογή, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας και την ιδιαιτερότητα των γεωγραφικών τοποθεσιών. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να λέμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και υποδομές στα λιμάνια για την ενέργεια, για τις μεταφορές που να είναι βιώσιμες και αηφόρες, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές. Όσον αφορά τον τουρισμό, και ξέρετε πόσο πολύ με ο τουρισμός, συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις του συναδέλφου. Όμως και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη επενδύσεων στο φυσικό μας κεφάλαιο, το κεφάλαιο της φυσικής μας κληρονομιάς και να φροντίσουμε για την αποκατάστασή του στις πρωτεύουσές μας. Και να προσφέρουμε και κατάρτιση προσαρμοσμένη και δεύματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί συχνά βλέπουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα και τίποτα. Και τελικά είναι η οικονομία αυτή που προέχει. Τώρα για τη θάλασσα. Η συνύπαρξη ανθρωπίνων ε, δραστηριοτήτων πρέπει και αυτή να εξεταστεί. Δεν πρέπει να έρχεται σε ανταγωνισμό. Μίλησες πριν για την αλία, για την υδατοκαλλιέργεια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες. Πρέπει δηλαδή την γαλάζια ανάπτυξη να τη συνδέσουμε επίσης και με την ασφάλεια στη θάλασσα, όπως επίσης και με την αρχή της προφύλαξης. Αυτά έχω να πω. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω, γιατί όπως είπα συμφωνώ απόλυτα με τα όσα ακούσαμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Δανέλη για την έκθεσή του. Μέχρι τώρα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά μαζί και στο μέλλον φαντάζομαι το ίδιο. Βεβαίως με ενθουσιάζει δε αυτή της γαλάζιας ανάπτυξης, την παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν σκεφτούμε ότι 70% της γης αποτελείται από νερό και 30% από γη και ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη του πληθυσμού στα επόμενα χρόνια, πληθυσμού ο οποίος θα θέλει και να φάει και να μεταφέρει προϊόντα και να ε, αποκομίσει ενέργεια από ενεργειακές πηγές που μπορεί να είναι και η θάλασσα, έχουμε πολύ μεγαλύτερο ρόλο να περιμένουμε να διαδραματίσει η θάλασσα στο μέλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να αναλογιστούμε αυτή η ανάπτυξη, πώς μπορεί να δημιουργηθεί, πώς μπορούμε όμως ταυτόχρονα και να προστατέψουμε τους ωκεανούς μας για την ανθρώπινη δραστηριότητα και από την ανθρώπινη δραστηριότητα και βέβαια πώς μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε κομμάτι αυτής της ανάπτυξης στο μέλλον. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Η γαλάζια ανάπτυξη είναι συμβολή πολύ πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Χρειαζόμαστε και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας που μπορούμε να δημιουργήσουμε στο χώρο της θάλασσας και βεβαίως ε, πια πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει του σαλονιού θα λέγαμε και η ε, πολιτική για τις θάλασσες γιατί στο παρελθόν θα θυμάστε ότι ήταν παραγωνισμένο ο ε, τώρα έχει και δική της γραμμή στον προϋπολογισμό, είναι πια κομμάτι της ευρωπαϊκής μας στρατηγικής και είναι πολύ σημαντικό αυτό τομείς του μέλλοντος επίσης βλέπω ότι αναφέρονται. Εμείς στη Γερμανία ε, είχαμε την διεθνή διάσκεψη για τις θάλασσες, στην οποία έλαβα μέρος και χωρίς να ονομαστεί με αυτό τον τίτλο ακριβώς, η γαλάζια ανάπτυξη είχε πολύ μεγάλη σημασία στην ε, συζητήση της διάσκεψης αυτής. Βεβαίως οι μεταφορές έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα έχουμε τα υπερπόντια ε, πλοία τα οποία θα ταξιδεύουν πολύ πιο συχνά πλέον στους ωκεανούς μας και άρα χρειάζονται και green shipping, πράσινα πλοία, πιο ασφαλή πλοία, πιο περιβαλλοντικά ε, πλοία, πιο οικολογικά πλοία. Βεβαίως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, την ενέργεια που μπορεί να μας προσφέρει η θάλασσα και η αιωλική ενέργεια και νομίζω ότι μπορούμε ε, και στις εγκαταστάσεις offshore να αξιοποιήσουμε αυτές τις πηγές ε, ενέργειας και να τις δώσουμε και σαν λύση μεταφορών. Σε μια διάσκεψη που είχαμε κάνει στη Γερμανία πριν από μερικά χρόνια, είχαμε την ευκαιρία να δούμε νέες εναλλακτικέ για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και την ενέργεια που προκύπτουν. Για τον τουρισμό επίσης, Βεβαίω όλοι προτιμάνε να πάνε στη θάλασσα, σχεδόν όλοι, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν, ε, να κάνουν τα μπάνια του το καλοκαίρι ε, ή να περνάνε τι διακοπέ του. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό. Μην ξεχνάμε και τον τουρισμό των πιο ηλικιωμένων τη τρίτη ηλικία. Το έχει εκθέσει πολύ ωραίο ο μα αυτό στην έκθεση. Ε, Ασφαλώς όμως χρειάζεται να υπάρχει και η προστασία του ε, θαλάσσιου περιβάλλοντος ε, από, και από τον τουρισμό εφόσον ε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες και σε σχέση με τις εγκαταστάσεις offshore και με τις αλληλευτικές εγκαταστάσεις. Για την αλληλεία. Είπαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για τις ηχθειοκαλλιέργειες σε απομακρυσμένες από τις ακτές περιοχές, offshore δηλαδή. Ε, αυτό είναι καλό, πρέπει να το αξιοποιήσουμε, δημιουργεί θέσει εργασία. Η γαλάζια βιοτεχνολογία που αναφέρεται επίσης, έχουμε ένα 10% ε, μόνο από τους ωκεανούς που αξιοποιείται ε, ως προς τα στοιχεία, ηχνοστοιχεία ή άλλα που μπορούν να προσφέρουν, αλλά και για τα φάρμακα και για τα καλλιντικά υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Υπάρχει τεράστιος πλούτος ωκεανούς που μπορούμε να αντλήσουμε. Βέβαια πάντα το πρόβλημα πάντα είναι οι μεταφορές. Βιοτεχνολογία λοιπόν πάλι εντάσσεται σε αυτή την ιδέα και ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουν στον καταναλωτή τα προϊόντα αυτά. Η εξόριξη από τις θάλασσες επίσης είναι πολύ σημαντικός ε, τομέας ε, να γίνεται ωστόσο με οικολογικούς τρόπους, με τρόπους οικονομικά σωστούς. Παρακολουθούμε την κατάσταση και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε και εγώ να πω ότι θα είμαι παρόν, παρούσα όταν υπάρξει εξέλιξη στο θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε βέβαια και τι αρμοδιότητε όπω υπόθηκε. Δεν θέλουμε να ε, γίνονται επικαλύψεις εργασιών και θα πρέπει στη στρατηγική μας να εμπλέξουμε τους, ε, όλους τους ενδιαφαρομένους, στρατηγική ε, σε σχέση με τρίτα κράτη, είπαμε και το θέμα της θεώρησης που θα μας απασχολήσει φαντάζομαι, και ο κανονισμός για το θαλάσσιο χώρο, δηλαδή το πώς ε, θα χαράξουμε ενδεχομένω ε, ρότες για τα πλοία, το πού μπορεί να γίνεται η αλευτική δραστηριότητα, το πώς θα εντοπιστεί ο τουριστικός, η τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά για να έχουμε μια καλή ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Δανέλη για αυτή την έκθεση που είναι ένα καλό σημείο κίνηση. Έχω να κάνω κάποια σχόλια. Θα ξεκινήσω από τον τουρισμό, καθώς η Επιτροπή μας Μεταφορών και Τουρισμού. Να μην ξεχνάμε τη συνέργεια ανάμεσα ε, στον ε, παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, πώς αυτό συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό όχι μόνο για τους πιθανούς αρνητικ... πιθανές αρνητικές συνέπειες τουρισμού στο περιβάλλον. Χρειαζόμαστε ένα γενικότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Και άρα η χωροταξία εν προκειμένου είναι στοιχείο κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να δοθεί λοιπόν προτεραιότητα στην προστασία της θαλάσσιας και παράκτης βιπικιλότητας και χρειάζονται νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες λαμβάνοντας ακριβώς αυτή την προτεραιότητα υπόψη. Και να μην σημαίνει το αντίθετο, Δηλαδή να προσπαθούμε να πιέσουμε, να, να, να ταιριάξει η οικονομική ανάπτυξη με την εξόριξη ε, πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ. Θα πρέπει να ιεραρχήσουν προτεραιότητες έχω το βασικό γνώμονα την προστασία των παράκτημων και θαλάσσιων περιοχών. Στην παράγραφο 10 της ε, έκθεσης σας μιλάτε για τις διαφορές που έχουν τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη ε, συστημάτων διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων ε, περιοχών. Χρειάζεται πραγματικά συνέπεια ε, στην εφαρμογή αυτών των στρατηγικών διαχείρισης. Για παράδειγμα, η Βρετανική κυβέρνηση εξετάζοντα αυτό το, θέμα τη ταυτοποίηση τέτοιων ζωνών, ενέκρινε έως τώρα 31 τέτοιες ζώνες, ενώ οι πυρογνώμονε μα, είχαν συστήσει 127. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε να πιέσουμε πολύ περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να φανούμε πιο Ευρωπαίοι, αν θέλετε, και εμείς αυτό το το ό,τι αφορά τις άλλες πτυχές της γαλάζιας ανάπτυξης, πράγματι, δίνει ένα δυναμικό στην γαλάζια ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το δυναμικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να το εκμεταλλευτούμε τον τρόπο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε για τι προτεραιότητε για την αλλαγή του κλίματο. Με την κατασκευή, με την αυπήγηση νέων και καλύτερων οικολογικών πλοίων και αυτό σε συνδυασμό με τις εργασία, είναι κάποιο από τους στόχους ε, τη Λευκής Βίβλου ε, για τον ευρωπαϊκό, ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Και αυτό ο στόχο του 50% της μεταφοράς από τις οδικέ στις θαλάσσιες και στι εθνικές μεταφορέ το 2050 είναι κάτι που πρέπει να μην ξεχνάμε. Επίση, θέλω να υπενθυμίσω τους νέους θετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την χρήση ε, κεφαλαίων κινδύνου, venture capital για τέτοιου είδους project, ώστε να εγγυηθούμε καλύτερες επενδύσεις. Χαιρετήσουμε επίσης τις νέες ιδέες σχετικά με την κατάρτιση, εκπαίδευση, ιδίως μας στα πλαίσια του μοντέλου Εράσμους, για να βρούμε νέες δεξιότητες που ακριβώς έρθουν να ταιριάξουν στις ανάγκες της μεγάλης Αναπτύξης. Τώρα έχω και κάποια ε, μη τόσο θετικά, μάλλον αρνητικά ε, να πω. Δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ε, την εξόρυξη μετάλλων από τη θάλασσα που να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγάλο, τεράστιο κίνδυνο, ιδίως σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σύνεση εν προκειμένου. Το είπε και η προλαλή σα. Όταν δούμε ακριβώς ε, τι σημαίνει οικολογικός πολιτισμός ε, και γαλάζια βιοτεχνολογία. Για μένα υπάρχουν ακόμα θέες ζώνες εν προκειμένου. Ε, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους ε, και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα σχόλια ε, εξ ονομάτως του κ. Βαντάλεν, που είναι ο Σκιώδης. Πρώτα απ' να ευχαριστήσουμε τον ε, εισηγητή για την ε, πρόδειλος, προδήλωση μάλλον πολύ καλή δουλειά που έκανε, τον ενθουσιασμό που δείχνει μέσα από το κείμενό του και περιμένουμε να δούμε το σχέδιο έκθεσης. Μπορούμε να πούμε ότι πολύ συχνά και τα κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν τα ωφέλη και τις θέσεις εργασίας που δίνουν το μέσο τουρισμού. Είναι πραγματικά μια τεράστια λυσίδα ε, εφοδιασμού εν προκειμένου και πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε σαν τη σταχτοπούτα της οικονομίας. Πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ, θεωρώ. Επίσης, ο Πίτερ ε, είναι της γνώμης ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι φιλόδοξη και αυτό που του αρέσει και μας αρέσει είναι ότι θέτει τα θέματα κλειδιά εν προκειμένου. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την ναυτιλία, για τα πλοία, αλλά μιλάμε και για τις μεταφορές, για τις θαλάσσιες, και τον αντίκτυπο στις οδικές και τις ιδρυτικές μεταφορές. Άρα αφορά την ε, βιομηχανία εν γέννη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη με τη θαλάσσια μας ιστορία και για να μπορέσουμε να χαράξουμε το μέλλον τη. Στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και θα θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι αντιμετωπίζεται το θέμα της ρήπανσης, γιατί και εμείς ερχόμαστε από νησί και οι εκθέσεις μας είναι πάμπολες που και μπορούν να επηρεαστούν πολύ αρνητικά αν κάτι πάει στραβά. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις πτυχές για να είμαστε σίγουροι. Στην ε, έκθεση για την θαλάσσια πολιτική έως το 2018 τίθεται το θέμα της ε, ρήπανση των πλοίων και ίσως ε, τα πλοία που ρηπαίνουν λιγότερο να πληρώνουν λιγότερο. Η χρήση λοιπόν ε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι κάτι ε, σημαντικό εν προκειμένου. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό ε, για την επίλυση προβλημάτων διεθνών όπω αυτό που είδαμε στη Σομαλία, στην Ιγυρία. Χρειάζεται λοιπόν διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση τη πειρατεία. Είναι όλα θέματα πάνω-πάνω ε, στην ε, ατζέντα μα γιατί θέλουμε μια ασφάλεια στην βιομηχανία αυτή. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όλε τι εθνικέ κυβερνήσει. Επίση, ο Σκιώδη θέλει να μην ξεχνάμε ότι προνόμιο των κρατών μελών είναι το θέμα τη χωρο... πολιτική χωροταξία και η συνεργασία εδώ είναι η καλύτερη λύση. Όμω εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει εθνική κυριαρχία ε, σε αυτό το τομέα. Και κλείνοντα τα σχόλιά του, θέτει και κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα και αναφέρεται σε κάποιες άλλες ανακοινώσεις τις οποίες έχει θίξει και ο εισηγητής. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι θερμά ε, τον εισηγητή, ε, τον ευχαριστούμε εξ του του και περιμένουμε την επόμενη συζήτηση του θέματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Σπύρο Δανέλη για την πρόταση που μας παρουσίασε. Τον ευχαριστώ και εγώ γιατί είναι μια πρόταση την οποία ασπάζομαι θεωρώ ότι έχει χρηθεί το σωστό πλαίσιο στην πρότασή σας. Θέλω και εγώ να συμβάλλω στη συζήτηση που θα μεταφραστεί και σε συγκεκριμένες τροπολογίες. Θέλω να ξεκινήσω από μια πρώτη σκέψη το σύστημα της παράκτιας ανάπτυξης και η νησιωτική ε, οπτική γωνία προκειμένου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον προγραμματισμό. Είμαστε στη στιγμή στο σύστημα Ευρώπη 2020 και αυτό, αυτή είναι η πηξίδα μας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Θέλουμε μία Ευρώπη οικονομικά αναπτυγμένη από όλες τις απόψεις. Και σίγουρα στο ιστορικό της δεν μπορεί να έχει κάποια βαρύδια, να έχει κάποιες περιοχές, όπως είναι οι παράκτης, οι περιοχές, που υπολείπονται πολύ σημαντικά σε σχέση με άλλες περιοχές Ευρώπης και δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν όπως και οι άλλες. Για να υπάρχει λοιπόν μία έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη που να μπορούν να συμμετέχουν όλοι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλύσουμε τα διεθνωτικά ελλείμματα, τα διθρωτικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν σε αυτές τις περιοχές να αποτεχθούν εξίσου. Σίγουρα θέλω να σας υπενθυμίσω και κάτι άλλο και να σας επισημάνω το εξή. Σε επίπεδο μεταφορών και του κόστου των μεταφορών, κάτι που ε, ουσιαστικά τιμωρεί, αν θέλετε να πω, την τις πλέον απομονωμένες περιοχές, κυρίως στα νησιά, είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε περαιτέρω. Να δώσω ένα παράδειγμα έτσι για να μιλάμε συγκεκριμένα ε, πράγματα. Μιλάμε για τα προβλήματα των πολιτών, έτσι δεν μιλάμε γενικά και όριστα για συστημικά προβλήματα. Ε, όταν έχουμε ένα όχημα που συνδέει τη Σαρδινία με την υπηρετική Ιταλία, ένα αυτοκίνητο για τρία άτομα στοιχίζει 800 ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν αυτόν το κόστος μεταφοράς για 120 ναυτικά μίλια που είναι η απόσταση από το νησί στη Βρετική ε, Ιταλία. Πώς λοιπόν λειτουργεί τόσο αρνητικά για τους ε, πολίτες, την κυκλοφορία των πολιτών και την ε, διακίνηση αγαθών. Σκεφτείτε λοιπόν για πόσα νησιά μιλάμε. Στη Σαρδινία έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτε. Σκεφτείτε την Κρήτη και άλλα νησιά. Μιλάμε συνολικά για 5-6 εκατομμύρια ανθρώπου στη Μεσόγειο και μόνο που α, είναι σε μειονεκτική θέση πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε άρρηκτα αυτό το θέμα με τη λειτουργία της ενίας αγοράς. Ένα άλλο σχετικό σημείο, πάλι μιλώ για διεθρωτικά στοιχεία, και αναφέρομαι στον τουρισμό. Και έναν ακόμη συστημικό περιορισμό είναι ο εποχικός χαρακτήρας του τουρισμού, δηλαδή μία περιοχή να λειτουργεί με μια οικονομία που δουλεύει μόνο τέσσερις μήνες το χρόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά, 4-5 μήνες, έτσι. Ε, σκεφτείτε ε, τα μεγάλα νησιά. Ενώ για άλλες περιοχές, ακόμη πιο μονομένες, μιλάμε για μια οικονομία που λειτουργεί έναν-δύο μήνες το χρόνο. Είναι πραγματικά παράλογο να περιμένουμε ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικούς. Εν μέρη, ο Σπύρος Δανέλης αναφέρει αναφέρθηκε σε αυτά τα αισθήματα που αναφέρομαι και εγώ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αφαιρθούν στο κείμενο. Θέλω να κάνω και εγώ κάποιε προτάσει με τροπολογίε που ελπίζω να λάβει υπόψη. Και κλείνοντα, Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια σκέψη ακόμη. Το νομικό μα σύστημα μα δίνει και εργαλεία, όπω είναι ο Τηλενικός κώδικα, για παράδειγμα, που στο άρθρο 151 ο κώδικα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ορίσουν ένα ε, εργαλείο που είναι οι ελεύθερες ζώνες που μπορεί να προταθεί ως εργαλείο για να ξεπεραστούν αυτά τα διθρωτικά προβλήματα με μια πλεονεκτική φορολογική πολιτική για να αντιμετωπιστούν λοιπόν τέτοια ζητήματα, προβλήματα και με τέτοιου είδου τρόπου, τέτοιε διευθετήσει αν θέλετε, που αν θέλετε ουσιαστικά είναι που έχουν πολύ λιγότερη αρνητική συνέπεια από ότι ε, μια μεγάλη παρέμβαση από την πολιτική συνοχής ή άλλε κοινωνικέ παρεμβάσει στι εθνικέ πολιτικέ των κρατών μελών. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αντίθετα, και κλείνω πρόεδρε, αντίθετα με αυτόν τον τρόπο, με αυτέ τι διευθυντησει μπορούμε μια άπαξ ε, και διαπαντό να επιτρέψουμε να λειτουργήσει πραγματικά ενιαία χώρα αν προκειμένου. Και όταν θα μπορούσαν και αυτές οι αγορές να συμβάλλουν οικονομικά ε, στην ανάπτυξη, θα καταλήξουμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Αυτό πιστεύω και θα μπορούμε να μιλούμε για Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως και να το εννοούμε μέχρι κεραία σε αυτόν τον όρο. Ευχαριστούμε. Θέλω κι εγώ να πω δύο λόγια, να ευχαριστήσω κι εγώ τον κύριο Δανέλη για την ε, έκθεσή του αυτή. Το μόνο που έχω να πω είναι να θυμόμαστε και τον Βορρά και τα ύδατα εκεί, τα ψυχρά ύδατα, όχι μόνο τα θερμά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Και βλέποντας τι γίνεται με τα κουραζιερόπλια και το σχετικό κλάδο, αυτό που με απασχολεί σε ορισμένες χώρες μέλη είναι ότι υπάρχει μια μονοπολιστική αντιμετώπιση. Πέρα από τη δικιά μου χώρα έχουμε προσωπικό από το Σαθάμπτον και αλλού. Πρέπει κανείς να προσέχει να μην καταλήγει με ένα λιμάνι το οποίο να συγκεντρώνει όλα τα κουρασγερόπλια. Πράγμα το οποίο συμβαίνει στη χώρα μου. κύριε Κουσία και εσείς είχατε κάτι να πείτε. Εντάξει, έχουμε καθυστερήσει εξαιτία του συναγερμού φιάσκο, τέλο πάντων, α μην το πω φιάσκο. Ε, μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο. Σα ακούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Δανέλη για την έκθεση. Είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερος για τα νησιά, βέβαια θα σημειώσω όχι μόνο τα νησιά του Νότου, για όλα τα νησιά της Ευρώπης. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία αποτελεί ένα βήμα προόδου, πιστεύω, προς μια γαλάζια οικονομία και προς την ανάπτυξη. Και εκπροσωπεί η πρόταση αυτή ε, μια ιδεώδη λύση για το πώς μπορούμε να προαγάγουμε την ανάπτυξη, κυρίως στον χώρο των θαλασσών. Η καινοτομία, ο δυναμισμός πρέπει να μας οθήσουν προς τα μπρος. Πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά και αυτού του τομέα, ο οποίος μπορεί να στεφθεί με επιτυχία εάν κάθε κράτος μέλος, κάθε θεσμικό όργανο και κάθε περιφέρεια μέχρι την πιο μικρή επιχείρηση συμμετάσχουν στην προσπάθεια και τον αγώνα αυτών. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βοηθήσουμε και εμείς ώστε να αξιοποιηθούν κατά τρόπο αηφόρο οι ακτές μας. Συζητούμε λοιπόν το δυναμικό ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, την ενέργεια που μπορούμε να αντλήσουμε από τη θάλασσα τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ηχθειοκαλλιέργειες που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πιστεύω ότι κάθε ξεχωριστή πρωτοβουλία πρέπει να υλοποιείται με διαβουλεύσεις ή μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των εμπλοκομένων φορέων η γαλάζια αυτή η στρατηγική για την ανάπτυξη έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τουρισμό, για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι και άλλα νησιά θα βοηθηθούν ώστε να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητες των οικονομιών τους. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στο, στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα νησιά που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση, δεν θα ε, αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. δε τα κουραζιερόπλια, τα ποντοποραπλία που ξέρουμε ότι θα ενισχυθεί η παρουσία τους, διωγγώνεται ο τομέας αυτός τα τελευταία χρόνια και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν τον αγαπητό συνάδελφο για την εκθέση αυτή και περιμένω με χαρά να συζητήσουμε όλα τα θέματα και διμερώς ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι νιώθουμε πως μας ενθαρρύνει η σημερινή συζήτηση και τόσα έχουμε δει μέχρι τώρα από το σχέδιο του εισηγητή σας. Αυτό που μας ενθαρρύνει μας λέει συγχρόνω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε την πολιτική στη θάλασσα και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέεται με αυτήν. Σίγουρα έχει τεράστια σημασία η θαλάσσια οικονομία και εξαιτία του μεγέθους της, αλλά και εξαιτία του δυναμισμού που διαθέτει για να προσφέρει νέα ανάπτυξη. Κάποια από τα στοιχεία που είναι σημαντικά να λάβουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για ανάπτυξη είναι να γίνεται και όσο γίνεται καλύτερη διαχείριση του δυναμισμού αυτού. Μας ενθαρρύνει επίσης αυτό που φαίνεται και στην έκθεση αλλά και από τα σχόλια που ακούσαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή στην οικονομία που εξετάζουμε και να μην εξετάζουμε τον κάθε κλάδο και τον τάδε, το κάθε τομέα χωριστά. Να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή, να υπάρχουν διασυνδέσεις που να δείχνουν ότι η θαλάσσια οικονομία δεν σημαίνει μόνο η παράκτια περιοχή, αλλά έχει επιπτώσεις και στην ενδοχώρα και σε άλλους οικονομικούς τομείς που απορρέουν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η θαλάσσια οικονομία αποτελείται και από τους παραδοσιακούς τομείς, που μπορεί να είναι τα ναυπηγείες, αλλά και από νέους τομείς. Όλοι αυτοί οι τομείς λοιπόν, οι παραδοσιακοί και οι νέοι, οδηγούν στην καινοτομία και στην έρευνα κάτι πολύ βασικό για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εκεί όπου έχουμε επενδύσει σε καινοτομία, εκεί όπου έχουμε επενδύσει σε τεχνολογία, οδηγούν σε αηφόρο ανάπτυξη. Και είναι ακριβώς εκεί που εμείς είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Άρα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας για το μέλλον. Ακούσαμε για τις δεξιότητες και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι δεξιότητες γιατί, γιατί πρώτον πρέπει να διατηρήσουμε τι δεξιότητε, τι παραδοσιακέ που ήδη υπάρχουν, αλλά πρέπει βέβαια να στραφούμε και προ το μέλλον, να δούμε πώ εξελίσσεται η οικονομία στη θάλασσα και να φροντίσουμε να αποκτήσουμε τις κατάλληλες δεξιότητες, είτε πρόκειται για την ενέργεια από τη θάλασσα, είτε πρόκειται για συνδυασμό δεξιοτήτων, προκειμένου να αναπτυχθούν διάφοροι τομείς της θάλασσας που είναι ζωτική σημασίας. Μην κοιτάμε δηλαδή μόνο τι έχουμε μέχρι τώρα, αλλά και τι χρειαζόμαστε για το μέλλον. και πού διατομιακή δουλειά μπορεί να λάβει η χώρα για να συνδυαστούν δεξιότητες. Για τον ε, τουρισμό στη θάλασσα, ε, ξέρετε ότι και εμείς δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό και θα ετοιμάσουμε μια ανακοίνωση προς τα τέλη της χρονιάς. Είναι και το ε, θέμα της ημερίδας που θα λάβει η χώρα στην Βαλέτα 21 και 22 Μαΐου στη Μάλτα. Όσον αφορά τι δατοκαλλιέργειες, όλοι συμφωνούμε για το ότι είναι και αυτό ένας τομέας που έχει μεγάλο δυναμικό μπροστά του και που θα πρέπει να αναπτυχθεί παρετέρω. Να προσφέρει δηλαδή στην βιομηχανία τροφίμων. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ βέβαια για να φροντίσουμε συγχρόνως για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα για την εξόριξη ορυκτών. Εδώ πρέπει φυσικά να προσέξουμε πολύ τι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του τομέα αυτού, ο οποίος αναπτύσσεται σε ολόκληρο, τον, σε τη γη. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να το προσέξουμε πολύ και να δούμε πόσο θα υπάρξει ανάπτυξη της εξόριξης στα ανοιχτά της θάλασσας, offshore. Αλλά θέλει πολύ προσοχή. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα προθεθεί ο τομέας αυτός και πώς θα εξελιχθεί παρετέρω. Σίγουρα αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί και πρέπει να γίνει μελέτη αντικτύπου για να δούμε τι δυνατότητες και τι ευκαιρίες μας προσφέρει ο κλάδος αυτός. Πάλι για την ολική ενέργεια αποτελεί στοιχείο κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και άλλοι βέβαια που έχουν μεγάλη σημασία στα πλαίσια της ανάπτυξης. Η γαλάζια βιοτεχνολογία τα αναφέρατε, δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ τίποτα. Μερικά πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα, η ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί πολύ από τις ε, γενικότερες προϋποθέσεις, από τις συνθήκε που θα προσφέρουμε, από το γενικό κλίμα που θα επικρατεί. Οι προτάσεις που υπάρχουν σήμερα έχουν να κάνουν με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα διαφορετικά ταμεία, λίγο πολύ πώς αλλιώς να το περιγράψω. Για την καλάζια ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτά να ακουστούν και να συζητηθούν στα κράτη-μέλη μεταξύ κρατών μελών και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να φροντίσουμε να αναπτυχθούν παρετέρω τέτοια προγράμματα γαλάζιας ανάπτυξης. Για την ε, ανάπτυξη της παράκτειας οικονομίας μεταξύ άλλων. Τα μέσα τα οποία εμείς προτείνουμε σαν ολοκληρωμένα εργαλεία είναι η γνώση, η επιθεώρηση και η θαλάσσια χωροταξία, χωροταξία του θαλάσσιου χώρου. Για μας αυτά τα τρία είναι αλληλένδετα και απαραίτητα για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας γνώση, γιατί όλοι χρειαζόμαστε δεδομένα και πρέπει να βασιζόμαστε σε δεδομένα, άρα χρειάζονται όλο και περισσότερα για να διευκολυθούν και οι οικονομικοί εταίροι. Έπειτα χρειαζόμαστε επιθεώρηση, γιατί χρειαζόμαστε ασφάλεια, χρειαζόμαστε βιωσιμότητα και θα, θα χαροταξία του θαλάσσιου χώρου, γιατί χρειαζόμαστε τι καλύτερε δυνατόν συνθήκε ώστε να μπορέσουν και οι οικονομικοί φορεί να δράσουν στη θάλασσα. Αυτά προ το παρόν, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κύριε Δανέλη, εσεί έχετε να προσθέσετε κάτι. Σύντομα όμω, σα παρακαλώ. Γιατί όπω είπαμε, χρειάστηκε να βγούμε πριν και μείναμε πίσω κάπω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η, εμπειρία που έχουμε ε, σε σχέση με τη θαλάσσια οικονομία και κυρίως βεβαίως με τον τουρισμό, τον παράκτιο και τον ε, νησιωτικό, αλλά και στους άλλους τομείς, ε, οι θετικές και αρνητικές γνώσεις μας ε, μας κάνει σοφότερους σήμερα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το βασικό κεφάλαιο το οποίο επενδύουμε όχι μονάχα στον τουρισμό αλλά στο σύνολο ε, των τομέων των αναπτυξιακών της γαλάζιας ανάπτυξης ε, είναι το περιβάλλον. Η, ποιότητα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του εξαιρετικά ευαίσθητου οικοσυστήματος του θαλάσσιου είναι κλειδί για την περαιτέρω ε, αναπτυξιακή διαδικασία στη θάλασσα. νομίζω ότι συμφωνούμε με, το, με την Επιτροπή και βεβαίως με τους συναδέλφους όλους για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια και τη συνεργασία τους. Ε, νομίζω ότι ε, ο, ο πιο αμφιλεγόμενος τομέας ε, είναι βεβαίως η εξόριξη των ορυκτών του βυθού της θάλασσας. Είναι ένας τομέας που είτε μας αρέσει είτε όχι. Επειδή είναι εξαιρετικά δυναμικός, έχει μία πορεία μπροστά του πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ιδιαίτερα και νομίζω ότι αυτό που ζητείτε είναι να βάλουμε από την αρχή σαφείς ε, και αυστηρούς κανόνες στο παιχνίδι και να μπορούμε να, τους, να ελέγχουμε αν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Ε, κλείνοντας θέλω να πω ότι ε, ό,τι λέμε ισχύει βεβαίως για το σύνολο των θαλασσών της ε, Ευρώπης, όχι μόνο για τη Μεσόγειο αλλά και τη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική κτλ και ε, να πω ότι τις επόμενες ημέρες ε, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία ε, να κατατεθούν οι τροπολογίες, οι προτάσεις για τις τροπολογίες από τους συναδέλφους θα έχουμε τη δυνατότητα για την, τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα διότι είναι πολλά τα ζητήματα που μπορούν να προσθεθούν αλλά η οικονομία του χώρου τον οποίο είχαμε στη διάθεσή μας δεν μας επέτρεψε να αναφερθούμε σε άλλα επιμέρους ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και ε, στην επόμενη φάση της συνεργασίας μας με χαρά. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Δανέλη. Προθεσμία 29 Απριλίου και ψηφίζουμε 30 Μαΐου. Επόμενο θέμα τώρα. Πάμε πίσω στον κύριο Σαρβάμα είναι η έκθεσή του για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Σρι Λάνκα. Συγγνώμη κύριε Σαρβάμα, αλλά μπλεχτήκαμε με τον συναγερμό και απλώς ξαναρχίσαμε μετά. Τώρα έχετε εσείς το λόγο για τη δικιά σας την έκθεση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Πρόκειται για ένα από αυτού, μια από αυτές τις ε, συμφωνίες που ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες αφορά την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, λαϊκή δημοκρατία της ε, Σρι Λάγκα. Ύστερα από τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Σρι με κάποια ευρωπαϊκά κράτη, προβλήματα δεν υπάρχουν. Ψηφοφορία προβλέπεται στα τέλη Μαΐου, αν δεν Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπένιεν. Ναι, Πρόεδρε, κερδίζουμε χρόνο νομίζω να πούμε ότι υποστηρίζουμε πλήρω ε, την πρόταση του συγητού και μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έτερος, Φώστερ παρακαλώ. Συμφωνούμε. Προθεσμία για κατάθεση πλήρως τροπολογιών και η μόνη τροπολογία μπορείτε να καταθέσετε είναι για απόρριψη 24 και ψηφοφορία Απριλίου και ψηφοφορία στις 7 Μαΐου. Ε, η Επιτροπή θέλει το λόγο, όχι ευχαριστώ. Και άρα πάμε στο τελευταίο θέμα της ημέρης της διάταξης, η έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου για την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Έχετε το λόγο κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Ήδη έχω προτείνει και εγώ κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Είχα επαφή με τους κοιόδους στο Στρασβούργο και πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία και για τις πιο πολλές τροπολογίες και τις συμβαστικές. Περιμένω την ψηφοφορία στην Επιτροπή Επασχόληση για τη γνωμοδότηση και μετά θα έρθω εδώ με τις τελευταίες συμβαστικές τροπολογίες και ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπένιεν. Ναι. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση μεταξύ των σκιώδων και του εισηγητή στο Στρασβούργο. Ε, οι πιο πολλοί συμβιβασμοί έχουν συμπεριλάβει τις και μου ήταν εξαιρετικά πραγματικά όλα και πρέπει να αναφερθούν ε, και οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι καταναλωτές. Αυτό ήθελα εγώ να είμαι σίγουρος, γιατί ε, υπάρχει και ένα συμφέρον των επιχειρήσεων εν προκειμένου. Επίσης, να βλέπω πολύ θετικά για το συμβασμό που υπέβαλε ο εισηγητής ε, για, ε, τους, για τα κομβικά αεροδρόμια, τα hub airports και για τα περιφερειακά αεροδρόμια και για την καλύτερη εξειδίκευση που κάνει σε σχέση με τις υποδομές. Ε, κάποια άλλα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί και ελπίζω να επιληθούν στο μέλλον είναι η τροπολογία 60 που υπέβαλα Είμαστε της γνώμης ότι η Κομισιόν δεν μπορεί απλά να ε, διευκρινίσει τα θέματα της συμμετοχής της Ένωσης στον ΙΚΑΟ, εν προκειμένου έχει λόγο το Συμβούλιο. Χρειάζεται μια, διε, μια διευκρίνηση, μια διόρθωση, ε, δεν ξέρω ακριβώς που να γίνει εδώ. Και για την τροπολόγια 54, Είχε συμφωνήσει πιστεύω ο εισηγητής με την προσέγγιση, δηλαδή χρειάζεται καλύτερη συνεργασία για να εγγυηθούμε την αποτελεσματική υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Δεν πιστεύω όμως ότι έχει θίξει ποιοι είναι οι πραγματικοί φταίχτε που ε, αποτελούν τροχοπέδι στο να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Ε, ελπίζω να έχει συμφωνεί με μια προφορική τροπολογία που θα υποβάλω. Κυρία Λιχτενπέργκερ, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία στη συνεδρία της στο Στρασβούργο. Θέλω να επισημάνω ότι το θέμα της συγχωρήπανσης ε, στα αεροδρόμια έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Το λέω γιατί υπάρχει και μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πρόκειται να επικαιροποιηθεί και ασκήθηκε πίεση προκειμένου να αρθούν κάποιοι κανόνες για αμερικανικά αεροπλάνα τα οποία θεωρούνται υπέτεια για την χορύπανση. Ε, πρέπει λοιπόν και το θέμα αυτό να το λάβουμε υπόψη το πλαίσιο των ευρωπαϊκών ενιαίων ευρωπαϊκών ουρανών είναι πιστεύω πολύ σημαντικό το ότι ακολουθεί μια σαφή γραμμή όσοι της ευχαριστώ κυρία Φώστερ ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαρινέσκο δεν χρειάστηκε δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα στο, στη συνεδρίαση γιατί ήμουν στο Ερωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία και τις συμβαστικές τροπολογίες όπως τις έχουμε δει. κάποιες σημεία ίσως ήθελα να τα δω χωριστά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο, το θέμα του υπερσιβηρικού με απασχολεί. Είναι σημαντικό Πρέπει να μιλήσουμε επίσης για το θέμα των επιπλέον, ε, του επιπλέον δυναμικού των αεροδρομίων για διαδρόμους και τα λοιπά, νέους διαδρόμους. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μαρινέσκου θα περιμένει και τη γνωμοδότηση Επιτροπής ε, Απασχόλησης πριν καταλήξει. Πάντως εν γέννη έχουμε μια σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σολχαντράουι. Ευχαριστώ αντικοθιστώ τον συνάδελφο Γιώργο Φλάχιτς, ο οποίο είναι στο εξωτερικό. Η ομάδα μου είναι ιδιαίτερα θετική. Πιστεύει ότι είναι ένα πολύ καλό κείμενο και στο Στρασβούργο συζητήσαμε. Οι σκιώδεις είχαν πολύ καλή συνάντηση. Όλες τις συμβαστικές μπορούμε να τις στηρίξουμε. Και χαιρόμαστε που ο συγκητής έχει αντιδράσει θετικά και έχει στηρίξει πολλές από τις δικές μας τροπολογίες. Και έτσι έχει συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Θέλω όμως να προσθέσω ότι για μας υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες κλειδί που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικές. Οι 17 και 18, οι 36 επίσης. Όσον αφορά τη 17 και 18, εδώ θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι αθέμητος ανταγωνισμός και μέσα στην Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να είμαστε δυνατοί και εκτός Ευρώπης. Γι' αυτό και πρέπει να αποφύγουμε αθέμητες πρακτικές από τις χαμηλού κόστου αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα, ή από ενισχύσεις που δίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Να μελετήσουμε λοιπόν αυτή την πτυχή. Όσον αφορά τροπολογία 36, εδώ υπάρχει διατύπωση για τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες για προδιαγραφές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές. Είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να συντονιστούν οι δράσεις μας. Για μας είναι το ελάχιστο προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον διεθνή ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή την εξαιρετική αυτή η εκθέση. Θέλω να τον συγχαρώ, όπως να συγχαρώ και τους ε, άλλους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου για τις ε, τροπολογίες που υπέβαλαν μεταξύ αυτών των τροπολογιών βλέπω ότι οι περισσότερες μπορούν να ενισχύσουν αυτό το σχέδιο έκθεσης και να στηρίξουν μια πιο φιλόδοξη εξωτερική πολιτική αεροπλοεία για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις ε, που έχουμε ε, ενώπιόν μας. Μια σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σίγουρα θα μας βοηθήσει στην εφαρμογή και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, αλλά και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έγινε μέσω της ανακοίνωσής μας. Αν συμφωνείτε, Πρόεδρε, κάνω τα σχόλια μου προς τον εισηγητή σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, ε, να μην τα κάνω όλα αυτά τα σχόλια εδώ λόγω του χρόνου. Απλά ήθελα να επισημάνω εδώ μόνο λίγα ε, πράγματα ε, που μας απασχολούν ιδιαίτερα και τα υπόλοιπα σχόλιά μας θα τα δώσω υπόψη του εισηγητή της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα η τροπολογία 9. Θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο έτσι να κτίθεται η Επιτροπή ότι έχει χάσει ευκαιρίες συναρμόνιση της νομοθεσίας. Αυτό το κάνουμε καθημερινά. Επιδιώκουμε συνεχώς την περαιτέρω εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τροπολογία 9 μάλλον δεν είναι πολύ ορθή. Τροπολογία 13 Και μια πρόταση να μιλήσουμε για τα κατάλληλα πρότυπα και όχι ψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά ε, την ε, ασφάλεια. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ε, προτείνει υποβάθμιση σε σχέση με αυτό που επιδιώκει η η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιδιώκει πάντα πολύ ψηλά πρότυπα. Τροπολογία 27. θεωρώ ότι δεν υποστηρίξει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής και απλά ζητά πιο ψηλή φορολόγηση του κλάδου, κάτι που θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προσκόμματα ε, στις ε, διεθνείς ε, αγορές. Τροπολογία 28 δεν μας είναι απόλυτα σαφές τι περιμένει, τι προσδοκάει η Επιτροπή σας από εμά. Μιλάει για α, εύκολα προσβάσιμες ε, μελέτες. μους θέλετε να τη δυνατότητα να εξετάσετε πιο στενά ε, θέματα νησοτήτων ε, σε ό,τι αφορά τέλη, φόρους κτλ. Έπειτα, 46. Καλείται η Επιτροπή να ε, προτείνει ελάχιστες δεσμευτικές, ε, μάλλον ελάχιστους δεσμευτικούς ε, κανόνες. Στις συμφωνίες που έχουν συνάψει τα κράτη-μέλη με τα κράτη, διμερείς συμφωνίες, αυτές ισχύουν και εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε άλλα ελάχιστα υποχρεωτικά πρότυπα που να υπερέχουν Μπορούμε να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να συμπεριλαμβάνουν κάποιε στανταρίτρε στι διμερεί συμφωνίε, όπω αντίστοιχε έτσι να υπάρχουν σε ευρωπαϊκέ ε, συμφωνίε με τι χώρε. Τροπολογία 38. Εμείς ε, προτείναμε την αναθεώρηση του κανονισμού 868 που αφορά τον αθήμα του ανταγωνισμού ανάμεσα ευρωπαϊκούς και μη ευρωπαϊκούς ε, Ε, καθώς ε, οι μη Ευρωπαίοι μεταφορές έχουν ένα αθέμητο πλονέκτημα λόγω κρατικών ισχύσεων κτλ. Ε, είμαστε δικασία επανεξέταση του κανονισμού αυτού. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε ταυτόχρονα και με την πρόταση για τους εναλλακτικές πολιτικές πολυτροπικές ε, μεταφορές. Αυτό αν εννοούμε ουσιαστικά τα καθαρά αυτοκίνητα, του σύνδρομου υψηλή ταχύτητα. Ναι. Υπάρχει όμως μια αντιστοιχία σε αυτά που συμβαίνουν και που συμβαίνουν στο κόλπο τη ΕΠΑ. Προσπαθούμε λοιπόν να καταλάβουμε ουσιαστικά τι είναι με αυτή την τροπολογία, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά εντάχει, Πρόεδρε. Έπειτα και τροπολογία 40. Λέτε εδώ ότι η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει με μία σειρά γειτονικέ χώρε μεταξύ αυτών και Αλγερία. Να σα ενημερώσω ότι ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσει με Αλγερία. Έχουμε λάβει εντολή, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει αυτέ τι διαπραγματεύσει. σω ε, είναι καλό να διορθώσετε αυτή την τροπολογία. Επιτροπολογία 59. Εδώ καλείται την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το θέμα πριν θεσπίσει τυχόν προς τις κυρώσεις που θα σημειώνουν την ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορέων. Πάντοτε με προσοχή προσπαθούμε να εξετάζουμε τα πράγματα και η ανακοίνωσή μα ήταν μια προσπάθεια να δείξει ότι μελετούμε με προσοχή τα βήματα που προτείνουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τα μέτρα μα να θεωρούνται κυρώσει, αλλά ότι είναι μάλλον μέτρα υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ομηχανία. Και τέλο για την τροπολογία 60. Η... Καλείται την Επιτροπή να προτείνει διαπραγματευτικές εντολές για να δημιουργηθεί η θέση μας ε, στην ΕΚΑΟ. Μα ήδη αυτό έχει γίνει από το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καμία θετική ανταπόκριση από το Συμβούλιο. Αν θέλετε ιδανικός πώς είναι καλή αυτή η πρόταση αλλά ακόμα και σήμερα θεωρούμε ότι δύσκολα θα τύχη α, υποστήριξης και δύσκολα θα εφαρμοστεί. Αυτά. Ευχαριστώ και πάλι ε, Πρόεδρε και συγχαρητήρια στον οδηγητή. Ευχαριστώ κύριε Μαστινέσκου. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Θα τα λάβω υπόψη μου. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. 5 μα ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας. Θέλω να υπενθυμίσω 7 Μαΐου είναι η πρώτη μέρα που θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε, αλλά ίσως τον Ιούνιο. Αυτά. Έτσι τελειώνουμε για σήμερα το πρωί. Και σας ευχαριστώ όλους για την βοήθειά σας που καταφέραμε να ξαναρχίσουμε. Θα τα ξαναπούμε στις 3.